σοβιετικά στα θέματα, αλλά ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία για την Ευρώπη και λόγω του βραβείου Νόμπελ είναι σημαντικό να θυμηθούμε και την εξέγερση της Ουγγαρίας του 1956. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Äh, Διαδικαστικά. Κύριε Ντεσιλβέστης, έχετε το λόγο. Μόνο πέντε δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε. Έστειλα πολλά email. Στείλατε πολλά email για τη φωτογραφία αυτό και είπατε ότι θα χρησιμοποιήσω